Θα ήθελα όλοι να προσέξετε σε αυτά τα οποία θα πω. Θα σας δώσω όμως ένα λεπτό για να προλάβετε να καθίσετε εν τω μεταξύ. Oh, Ε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Αναφερθώ σε δύο συμβάντα τα οποία συνέβησαν εν πάση πριν λίγες μέρες και πρέπει να εκφράσουμε την κατανόησή μας την Παρασκευή στις 30 Οκτωβρίου έσπασε μια φοβερή πυρκαγιά σε ένα κλαμπ στην, ε, στο Βουκουρέστι όπου είχαν μαζευτεί 400 σχεδόν νέοι άνθρωποι. Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 46 μέχρι τώρα και άλλοι 100 βρίσκονται στο νοσοκομείο, πολλοί από αυτούς σε πολύ κακή κατάσταση. Οι σκέψει μας λοιπόν είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Ταυτόχρονα ακούσαμε με μεγάλη θλίψη την πτώση του ρωσικού αεροσκάφους, το οποίο προκάλεσε το θάνατο 224 ατόμων και εδώ πάλι ε, οι σκέψεις μας βρίσκονται με τις οικογένειες των θυμάτων. Κύριε Νεγκρέσκο, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, πήρα το λόγο γιατί ήμουν αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με άλλους Ρουμάνους βουλευτές να αναφερθούμε στον θάνατο των 50 αυτών ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην δισκοτέκ του Βουκουρεστίου. Πρόκειται για νέους ανθρώπους αγγεδμένα στη ηλικιακά Πολλοί από αυτούς παλεύουν, δίνουν αγώνα για τη ζωή τους και πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε μια δύσκολη περίοδο ε, για την χώρα μου. Ευχαριστώ τις διάφορες χώρες που ζήτησαν και προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν.